για τα θέματα αλλιές. Πριν περάσω στο επόμενο θέμα πρέπει να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ε, ε, μου ε, ανακοίνωσαν τον ορισμό της κυρίας Ανέτ Κόβιους αντικαταστώντας τον κύριο Λένε. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 4, παράγραφος 1 και 4 του κανονισμού, λαμβάνουμε υπόψη μας την εκλογή της κυρίας Ανέτα Κοέβιους από τις 12 Μαρτίου του 2014. Καλωσορίζω τη νέα συνάδελφο και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, πριν από τον έλεγχο των διαπιστευτηρίων της, η κυρία Κοέβιους παίρνει τη θέση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την προϋπόθεση ότι έχει κάνει την δήλωση ότι δεν ασκεί μια άλλη δραστηριότητα ασύμβατη με αυτή του Ευρωβουλευτή. Πήρα επίσης από την ομάδα Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τις αιτήσει για τη συμμετοχή της κυρίας Κοέβιους στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων